κύριε, το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση Schwab για τις ε, παραβάσεις του ε, δικαίου ανταγωνισμού. Να δώσουμε πρώτα το λόγο στον κύριο Schwab. Ευχαριστώ τα μάλα κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Μάσο, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφέρω θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Αντιπρόεδρο κύριο Αλμούνια για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε για το θέμα αυτό. Αλλά κύριε Μάλσομ και εσείς μια χαρά είσαστε. Πολύ χαίρομαι για την παρουσία σας γιατί και εσείς έχετε συνεργαστεί πάρα πολύ θετικά με το Κοινοβούλιο και εμείς ήμασταν πολύ ικανοποιημένοι με όλα τα μέλη τη Κομισιόν και επίση και τον κύριο Κούρκουλα θα ήθελα χαιρετήσω ως εκπρόσωπο της ελληνικής προεδρίας και να τον ευχαριστήσω για τη δική του συμμετοχή στη διεκπαιρέωση αυτού του θέματος. Σε τελική ανάλυση όμως ήταν πάρα πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βρεθεί μια λύση και να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα να υπάρχουν ιδιωτικές προσφυγές κατά τον καρτέλ. Ο κύριος Σάτσε Περσέδο, ο κύριος Έπικ, ο κύριος Όλε Σμιτ, και η προκάτοχός του, επίσης ο κύριος ε, Μπασάικο και ο κύριος Ραπκάη έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Επίσης η επικεφαλής της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων λειτουργήσε και αυτή πάρα πολύ για τα θέματα αυτά. Εμείς επιτύχαμε τα θύματα των καρτέλ να μπορούν μετά από την εφαρμογή αυτής της οδηγίας να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους αν έχουν υποστεί μία ζημία και να μπορούν να καταθέτουν αγωγές στα δικαστήρια των κρατών μελών. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόοδος και θα πρέπει να την τονίσουμε ιδιαίτερα γιατί ακολουθεί την γραμμή που έχει χαράξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση για τον ανταγωνισμό της Ευρωπαϊκής Κομισιόν ότι πρέπει να υπάρχουν λεγόμενες δράσεις follow-on, οι οποίες ακολουθούν από μία απόφαση και επομένως με τον τρόπο αυτό να ξεπεράσουμε τους ε, κινδύνους να έχουμε αμερικανικού χαρακτήρα συστήματα συλλογικών αγωγών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πρόκειται μόναχα για την Κομισιόν, αλλά και για του συναδέλφου του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θέλω να αποτίσω φόρο τιμή, γιατί καταφέραμε να πετύχουμε να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξουν στρεβλέ εξελίξει όπω αυτέ που είδαμε στι Ηνωμένε Πολιτείε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα μπορέσουν να περάσουν από τον Ατλαντικό. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία παίζουν ένα ρόλο για τα θέματα αυτά, όχι μονάχα με την. Ε, ε δράση της Επιτροπής μας γιατί κάναμε πάρα πολύ σημαντικό, κάναμε πάρα πολύ σαφές ότι η αρχή μας θα πρέπει να είναι ότι θα πρέπει να μην γίνεται δεκτή η παραβίαση συλλογικών δικαιωμάτων. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία όπου θα μπορούσαν να υπάρχουν πρόοδοι και υπήρξαν πραγματικά βελτιώσει σε σχέση με την πρόταση τη Κομισιόν. Η σχέση μεταξύ του άρθρου 12 και του άρθρου 13, δηλαδή το ερώτημα ποια προνομιακή σχέση μπορεί να έχει κάποιος έναντι ενός καρτέλ, έχει καταφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θεσπίσει μια λογική ε, ρύθμιση και να περιορίσει αυτά τα δικαιώματα. Μπορεί λοιπόν μια προνομιακή σχέση με τον, ε, ε, για τον καταγγέλλοντα μπορεί να οδηγήσει στο να διαλευκαθούν καταστάσεις και να αντιμετωπιστούν παραβιάσεις του ανταγωνισμού. Κάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν για την Ευρώπη και καταδεικνύει και στι ΗΠΑ ότι δεν χρειάζεται κανεί να δίνει τόσα πολλά λεφτά για δικαστικού αγώνε. Μπορούν τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν πιο επωφελώ σε έρευνα και ανάπτυξη και τελικά με τον Τρίλογο καταφέραμε να εγκρίνουμε αυτή την άποψη η οποία είναι πολύ για την Ευρώπη. Και κατά δεύτερο λόγο, κύριε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε καταλήξει και σε ένα μηχανισμό για αντιστάθμιση ζημιών με εθελοντικό τρόπο και αυτό είναι πάρα πολύ θεματικό και κλείνω κύριε Πρόεδρε με τον τρόπο αυτό δίνεται μια ευνοϊκή δυνατότητα και στον καταγγέλλοντα να μπορέσει να αποκομίσει ε, αποζημίωση για τις ζημίες που έχει υποστεί χωρίς να καταφύγει στα δικαστήρια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Επίτροπο Μάλστρομ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρου αντιπροέδρου, του Αντιπρόεδρου Αλμούνια θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σβάμπ για τη δουλειά που έκανε, αλλά και τον κύριο Ράπκαη και τον πρόεδρο της Επιτροπής ΕΚΟΝ, την κυρία Μπόλτσα, και όλους τους κοιόδους συζητητέ και όλου όλους όσους επλάκησαν σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα της οδηγία ε, και την επικοδομητική στάση που είχατε. Μετά την επικοδομητική συνεργασία και των τριών θεσμικών οργάνων, η Κομισιόν πιστεύει ότι έχουμε φτάσει σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Καλωσορίζουμε, αλλά δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε σήμερα αυτή την οδηγία λίγο πριν διαλυθεί το Κοινοβούλιο, αλλά καλωσορίζουμε τα αποτέλεσμα της συνεργασίας. Ε, ο τύπος είπε ότι η οδηγία αυτή είναι η πιο σημαντική εξέλιξη στην πολιτική ανταγωνισμού τελευταία χρόνια. Ε, εκδημοκρατίζεται το δίκαιο ανταγωνισμού. Ο αντιπρόεδρο Αλμούνια είχε έρθει εδώ στην Ακρόαση πριν από τέσσερα χρόνια και σα υποσχέθηκε ότι το Κοινοβούλιο θα εμπλακεί πλήρω ε, σε αυτό το θέμα ως νομοθέτης. Και ως συνέπεια σήμερα ε, φέρνουμε αυτό το φάκελο που το διαπραγματευθήκαμε με την συνήθινη νομοθετική διαδικασία σε αίσιο τέλος. Ε, το δικαστήριο πριν από χρόνια αναγνώρισε ότι οποιοδήποτε θύμα είχε το δικαίωμα στην αποζημίωση. Αλλά στην πράξη ήταν δύσκολο να εξασφαλίσει τα δικαιώματά του. Πολύ λίγε αγωγέ είχαν γίνει οι καταναλωτές, οι μικρές επιχειρήσεις ε, με δυσκολία ε, εξασφάλιζαν αποζημίωση για την ζημία που υπέστησαν. Αυτή η οδηγία είναι ε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο πολύ σημαντική. Επιτρέπει στους πολίτες και στους επιχειρηματίες που έχουν φυγεί λόγω των δράσεων των, των, των καρτέλ να αναζητήσουν αποζημίωση. Ε, τα θύματα έχουν ε, δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στα αποδεικτικά στοιχεία για να στηρίξουν την ε, αγωγή τους. Ένας τρόπος για να τα εξασφαλίσουμε τα το δίκαιο των θυμάτων είναι να χρησιμοποιήσουμε το δίκαιο ανταγωνισμού. Επίσης, ξεκαθαρίζει τη σχέση μεταξύ το... του για την πρόσβαση των κειμένων. Το κείμενο που θα ψηφίσετε αύριο ε, δίνει κίνητρα σε εταιρείε να συνεργαστούν με τι αρχέ ανταγωνισμού μέσα των προγραμμάτων ευνοϊκή μεταχείριση. Να, αν ε, λειτουργούν αποτελεσματικά οι αρχέ ανταγωνισμού, είναι πολύ καλά νέα για τα θύματα ε, Όσο πιο αποτελεσματικά λειτουργούν οι αρχέ, τόσο πιο εύκολο θα είναι για τα θύματα να ζητήσουν αποζημίωση. Πετύχαμε σωστή ισορροπία. Από τη μία θα είναι πιο εύκολο τα θύματα να ασκήσουν τα δικαίωματα προ αποζημίωση και από την άλλη εξασφαλίζουμε ότι θα εφαρμοστεί σωστά ε, το δίκαιο ανταγωνισμού από τι αρχέ ανταγωνισμού. Και γι' αυτό σα ευχαριστώ όλου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ, Επίτροπε. Ο πρώτο ομιλητή είναι η κυρία Πέλτς για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή, τον κύριο Σφάπ. Αγαπητά μέλη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλά κράτη-μέλη αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά προσκόμματα για τους καταναλωτές και τους επιχειρηματίες, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, που είναι ε, δύσκολο να δικαιωθούν απολάβουν δικαιωμάτων που χάνουν όταν προβάλλουν αίτημα αποζημίωσης μέσα στα πλαίσια του δικαίου ανταγωνισμού. Σήμερα το θέμα είναι ύψη της σημασίας, δηλαδή να αρθούν αυτά τα προσκόμματα. Η όλη διαδικασία άρχισε εδώ και εννέα χρόνια. Ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία, χαίρομαι όμως διότι τώρα πλέον φτάσαμε σε αίσια αποτελέσματα. Πολλοί ε, συμμετείχαν στην όλη εργασία, ο κύριος Φαμπ και άλλοι συνάδελφοι, οι οποίοι ήταν πολύ αποτελεσματικοί στην εργασία αυτή και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να αποτίσω φορά την χορδμή στον κύριο Φαμπ για αυτή την εργασία. Τον συγχαίρω διότι αυτή είναι ευκαιρία, μια ευκαιρία για μας και για όλα τα ε, θύματα και τους καταγγέλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβάλλονται τα ε, δικαιώματά τους και προβάλλουμε αυτό το κεκτημένο μέσα στα πλαίσια μιας ρύθμισης, γενικότερης ρύθμισης και όχι υπερρύθμισης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε κατά πόσο έχουμε μία σωστή βάση για τη μελλοντική μας εργασία. Ε, η συλλογική αποκατάσταση έχει ε, ληφθεί υπόψη, καθώς και η πρόσβαση σε αποδεικτικά στοιχεία. Όλα αυτά τα ζητήματα τα έχουμε δει. Η πρόταση αυτή είναι εξισορροπημένη. Μιλάμε για μια εξισορροπημένη κατάσταση και για τον καταγγέλλοντα και για τον εναγόμενο και θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν, δεν θα υπάρξουν καταχρήσεις για αυτούς που θέλουν να προβάλλουν τα δικαιώματά τους για αποζημίωση. Δεν υπάρχει επίσης υπερβολική ε, ρύθμιση, δηλαδή υπερβολική γραφειοκρατία, έτσι ώστε να μην δοθούν υπερβολικά κίνητρα, έτσι ώστε οι καταγγελίες να είναι πολύ συχνές και άσκοπες. Επίσης, έχουμε βασιστεί σε μια γενικότερη συνένεση και όσον αφορά τις ε, αρχές, εάν προβάλλεται ένα επαρκές πλαίσιο αποζημίωσης, τότε θα ληφθεί υπόψη αυτό το πλαίσιο κατά την καταβολή της. Γνωρίζουμε ότι πολλές φορές υπήρχε θέμα χρόνου για τους καταγγέλλοντες και θεωρώ ότι ένας χρόνος είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Μιλάμε για κοινή εργασία που θα πρέπει να προβληθεί σε εθνικό επίπεδο. Ο κύριος ε, Σάντσος Πρεσέδο έχει το λόγο. Ως εισηγητής ε, της ε, πράσινης βίβλου μέσα στα πλαίσια του δικαίου ανταγωνισμού ε, καταφέραμε να εγκριθεί ένα ψήφισμα εδώ και 7 χρόνια και τότε ως εισηγητής είχα εκφράσει την ικανοποίησή μου διότι μιλούσαμε για μια πρωτοβουλία νομοθετικού περιεχομένου μέσα στα πλαίσια ενός τριμερούς διαλόγου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σφάμπ και τον κύριο Ραπκάη. Θα ενισχύσουμε τη, τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών μέσα στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς. Αυτά μέσα στα πλαίσια του δικαίου ανταγωνισμού που αποτελεί μέρος του DNA της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη συνθήκη της Ρώμης και ε, μετέπειτα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς οι αρμόδιες αρχές ε, δραούν έτσι ώστε να προβάλλουν ένα αποτρεπτικό χαρακτήρα σε απορριθμίσεις και ανισορροπίες. Μέχρι τώρα η κοινοτική πολιτική ανταγωνισμού τι έκανε προσπαθούσε να στυλιτεύσει τους, ε, τους εναγόμενους, ενώ αυτό που προσπαθεί τώρα πλέον να κάνει είναι να προστατεύσει τον πολίτη, τους ε, καταναλωτές. Δηλαδή μιλάμε για μια πρωτοβουλία η οποία προβάλλει την πεμπτουσία του δικαίου του ανταγωνισμού. Ο κύριος Αλμούνια κατά την ακρόαση πριν από το διορισμό του είχε αναφερθεί σε αυτό το ζήτημα. Πρόκειται για ζητήματα που σχετίζονται με την ε, νομική εποπτεία μέσα στα πλαίσια των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, προσπαθούμε να εξεύρουμε τρόπους έτσι ώστε να αποφύγουμε την ανασφάλεια δικαίου και να εξεύρουμε ε, λύσεις και εξοδικαστικά. Μιλάμε για καταγγελία και δυνατότητα δικαίωσης, δηλαδή αποζημίωσης, αλλά όχι υπερβολικής ε, αποζημίωσης. Έτσι υπάρχει πρόσβαση στα αποδεικτικά στοιχεία και αυτή η δυνατότητα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί βεβαίως αδικαιολόγητα και αυθαίρετα. Οι ιδιωτικές και αρμόδιες αρχές θα λάβουν υπόψη αυτή την δυνατότητα πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα έτσι ώστε οι αντισταθμίσεις να καταβληθούν μέσα στα πλαίσια του γενικότερου ορισμού των κυρώσεων. Έτσι προβάλλουμε και την αρχή της ε, χάριτος εκεί που μπορεί πραγματικά να προβληθεί μέσα στα πλαίσια του, της μεταχείρισης των ε, ΜΜΕ. Μιλάμε για τη δυνατότητα passing on και της δυνατότητας της Κομισιόν να δράσει άμεσα και ως μεσολαβητής. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν των μικρών παραπτωμάτων μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ε, τις αποζημιώσεις σε ένα ξεχωριστό πλαίσιο. Θα πρέπει λοιπόν, και όπως είδαμε τα δέκα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να συνεργαστούμε και σας ευχαριστώ πολύ ε, γιατί ήταν μεγάλη ικανοποίηση για ε, να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μία Ευρώπη μέσα στα πλαίσια της γενικότερης πρόοδου σε αυτό το ζήτημα. Eichhout. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι κλασικό ευρωπαϊκό θέμα αυτό και είναι και η σχεδόν η αίθουσα, ενώ το θέμα το οποίο συζητάμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε για τη δημιουργία συμπράξεων, καρτέλ, και αυτό μπορεί να έχει επιρροή σε πάρα πολλού ε, καταναλωτέ και μικρομεσαίε επιχειρήσει. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό αυτή η νομοθεσία να φροντίσει προκειμένου ο καταναλωτής και η μικρομεσαία επιχείρηση να μπορούν να αποζημιώνονται καλύτερα από τις ζημιές που δημιουργούνται από την δημιουργία συμπράξεων. Αυτό λοιπόν θα αγγίξει κάθε καταναλωτή και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σφάπ για τη συνεργασία γιατί σε κάποιες περιπτώσεις η συνεργασία, οι συζητήσεις ήταν πάρα πολύ έντονες αλλά τελικά ήταν πολύ καλή η διαδικασία και πετύχαμε μια καλή ισορροπία. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Σφάπ για την πολύ καλή συνεργασία. Είμαστε πολύ σκληροί από το περιεχομένου, αλλά πολύ ήπιοι με τις προσωπικότητες. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την καλή νομοθεσία. Να ευχαριστήσω και τους κοιότητες συζητητέ που κατέληξαν σε μια νομοθεσία που έχει ως σκοπό να προστατεύσει τον καταναλωτή. Επίση είναι σημαντικό γιατί αυτοί που θέλουν τελικά να καταγγείλουν τι συμπράξει, τα καρτέλ, με την νομοθεσία αυτή αντιευκολύνονται, γιατί η δάλο είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαρτυρήσει κανείς κατά μένος καρτέλ, γιατί συχνά προβάλλεται κανείς και ε, εκτίθεται. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το φροντίζει την νομοθεσία. Καλή ισορροπία, είμαι ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα. Φυσικά θα θέλαμε να είχαν ληφθεί και άλλα βήματα για τις συλλογικέ αγωγές για το collective redress. Ε, δεν θα εκπλήξει κανέναν αυτό και σίγουρα όχι τον κύριο Σφαμπ αλλά θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα πρώτο βήμα και προσβλέπω να συνεχίσουμε την επόμενη θητεία την ε, συζήτηση αυτή και με τον κύριο Σφάβο ελπίζω για τις λογική, συλλογικές συμβάσεις, ε, τις συλλογικές αγωγές. Ευχαριστώ. Η κυρία Τόμαζίτς, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Υποστηρίζω αυτή την πρόταση γιατί οι στόχοι είναι απαραίτητε προποθέσει για την δημιουργία μια κοινή αγορά και μια ελεύθερη κοινή αγορά. Ένα από του βασικού σκοπού τη κοινότητα αυτή. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα προκειμένου να εφαρμοστεί αυτή η καλή οδηγία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα των δικαστικών συστημάτων στα κράτη-μέλη, αλλά και ισορροπημένο επιχειρησιακό κλίμα όπου οι παραβιάσεις του δικαίου της περιανταγωνισμού θα τιμωρούνται και δεν θα αποτελούν καθημερινότητα. Δυστυχώς βλέπω ότι σε κάποια κράτη-μέλη αυτές οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται. Άρα, θεωρώ ότι θα μείνει κενή ε, περιεχομένου αυτή η καλή οδηγία. Η δική μου χώρα είναι μία από αυτές που το πολιτικό κατεστημένο υποστηρίζει τις μεγάλες επιχειρήσεις και καταπιέζει τις μικρές, οι οποίες διαρκώς ε, υπόκειται πιέσεις. Αυτό δεν γίνεται κατά λάθος, κατά τύχη. Είναι πολιτική. Η δικαστική λοιπόν μεταρρύθμιση είναι προϋπόθεση για σωστή καταπολέμηση της διαφθοράς και ε, εντάλλως θα συνεχίσουν να υπάρχουν παραβιάσεις ε, σε ό,τι αφορά την νομοθεσία τη αγορά. Θα υποστηρίξω το κείμενο αυτό, αλλά από κάπου θα πρέπει να ξεκινήσουμε, εν πάση περιπτώσει, να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Άντερ Στότερ, από ό,τι βλέπω, λέει ο πρόεδρος, δεν είναι εδώ. Και έτσι μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία Catch the Eye. Πρώτος ομιλητή, ο κύριο Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να τον κύριο Αλμούνια και τους άλλους επιτρόπους για το έργο τους τα τελευταία χρόνια στον τομέα. Δεν επενώ συχνά, όμως ο συναδελφός μου, ο Σουάμπ, αξίζει επένων. Θα ήθελα κάτι να κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσει να δουλεύει στον τομέα και γενικότερα στον τομέα του δικαίου ανταγωνισμού. Πολλοί πιστεύουν ορθώς, θεωρώ, ότι συμβαίνουν αδικίες και οι δικούμενοι δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν. Ας τους δώσουμε λοιπόν μια ευκαιρία να κάνουν κάτι. Είτε στο δικαστήριο, είτε εκτό δικαστηρίων. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τελευταίο ομιλητή. Κατά τη διάρκεια του κύριο Στολόγια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντική η έκθεση και θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσους συνεισέφεραν. Θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σε δύο σημεία. Καταρχήν χρειάζεται πιο στενή συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Κομισιών καθώς και κρατών μελών διότι θα πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο με το ανταγωνισμό διότι ο πρώτος κανόνας μιας σωστής αγοράς είναι ο κανόνας του θεμητού ανταγωνισμού και δίκαιου ανταγωνισμού. Επίσης, ε, στον τομέα της ενέργειας, του φυσικού, του φυσικού αερίου και ούτω καθεξής, ε, αν ε, σε ένα κράτος μέλος δεν υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός, τότε το, η διεθνής αγορά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επέβαλαν συγκεκριμένα σε μία χώρα να εφαρμόσει το δίκαιο ανταγωνισμού. Αλλιώς δεν μπορούσε να δράσει στην αγορά. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, συνάδελφε Στολογιάν. Και τώρα ολοκληρώθηκε λοιπόν η διαδικασία ΚΑΤΣΔΙΑ και τώρα θα δώσω το λόγο στην ε, Επίτροπο Μάλιμστρομ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, πολύ σύντομη αλλά και πολύ ξεκάθαρη και διευκρινιστική συζήτηση. Θα ήθελα να τα διαβιβάσω όλα αυτά στον Αντιπρόεδρο Αλμούνια, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορούσε να παραπληθεί μαζί μας σήμερα. Το τελικό κείμενο επί το οποίο συμφωνήσαμε είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για όλα τα θύματα των παραβιάσεων του δικαίου του ανταγωνισμού οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι καταναλωτές θα μπορέσουν να ε, γύρουν αξιώσεις ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Και επιπλέον το δικαίωμα αποζημίωσης θα ισχύει για τα θύματα που έχουν υποστεί πραγματικά τη ζημία και τα θύματα που δεν ε, είχαν άμεση σχέση με την παραβίαση επειδή ήταν πιο χαμηλά στην αλυσίδα και αυτό ισχύει συχνά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να πω ότι μιλάμε για πλήρη και δίκαιη αποζημίωση. Όλοι πιστεύουμε και υποστηρίζουμε ότι θα πρέπει να αποφύγουμε την πολλαπλή αποζημίωση. Εκ το κείμενο ρυθμίζει την διάδραση μεταξύ της δημόσιας και ιδιωτικής εφαρμογής του σχετικού δικαίου ανταγωνιστικότητα. Και τα προγράμματα ε, ε, λαμβάνονται υπόψη, επιμένοντας όμως στα, στις ψυχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των θυμάτων και σε θέματα διαφάνεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Σβάμπ, ευχαριστώ και τους ε, συνεισηγητές, τον κύριο Ραπκάι, την κυρία Μπόγλους και τους υπόλοιπους για την εξαιρετική τους εργασία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε Μάλμστρομ. Και τέλος, το λόγο έχει πάλι ο εισηγητής για δύο λεπτά, ο κύριος Σφάμπ. Καταρχάς να ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε, κύριε Βίλαντ, το γεγονός ότι έχουμε την ε, χαρά εδώ σήμερα. Δεν ε, είναι εδώ ο κύριος Αλμούνια. Χαίρομαι που είσαστε εσείς εδώ πέρα κύριε Μάλμστρομ και να πω ότι ακούσαμε αρκετά σε ευχαριστίες και χαίρομαι γι' αυτό, αλλά το θέμα είναι τα θέματα περιεχομένου. Και εδώ θα πρέπει να επανέλθω στο Σάντσο Εσπρεζίντο, να τον ευχαριστήσω γιατί ήταν πραγματικά και πολύ ευχάριστο στη συνεργασία και πολύ αποτελεσματικό. Θα μου λείψει πολύ. Και το ίδιο ισχύει και για τον ε, συνάδελφο Eichhout, αλλά κυρία Επίτροπε, αυτό που παραμένει ως εντύπωση στην οδογία αυτή είναι κάποιες ε, δεξιές ε, αμφιβολίες. Η απόφαση για το γεγονό, για παράδειγμα, ότι ο μάρτυρας ε, ε, παραμένει σε καθεστώς ε, θετικής μεταχείρισης και ευνοϊκής μεταχείρισης, για μένα θεωρώ ότι δεν είναι λογικό. Γιατί ο κίνδυνος που ενέχεται είναι κάτι το οποίο δεν κατανοώ γιατί τον διατρέχουμε. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μεγάλη πίεση προσπάθησε το άρθρο 11 να το συμπεριλήβει και ξέρω ότι πολλές αρχές στα κράτη-μέλη που ποτέ δεν είχαν κάποιον τέτοιο βασικό μάρτυρα τώρα έχουν ελπίδα και λάμπουν τα μάτια τους. Αλλά να μην μπλεκόμαστε. Το θέμα είναι να κατά πόσον υπάρχει επαρκής οικονομική δραστηριότητα και όχι το θέμα των μαρτύρων. Θα πρέπει λοιπόν τα επέμενα πόντε χρόνια να κοιτάξουμε το πώς θα δημορφωθεί αυτή η οδηγία και αυτό θεωρώ ότι θα οδηγήσει σε μια δίκαιη λύση τελικά. Αυτό που με χαροποιεί κυρία Αντιπρόεδρε Βίλαντ είναι ότι να εξαιρεθούν τα και απαντήσεων από την ε, οδηγία αυτή και να υπάρχει ένα ασφαλές περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και κυρίως να υπάρχουν καλύτεροι όροι για τους καταναλωτές. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι με ομοφωνία θα πρέπει να επιψηφίσει το σχέδιο αυτό, την έκθεση αυτή αύριο την ευχαριστώ πάρα πολύ λέει ο Πρόεδρος και έτσι ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Αύριο θα ψηφίσουμε στις 12 το μεσημέρι. Επόμενο θέμα είναι η έκθεση της κυρίας Ροδικράστας Ευεροπούλου σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια. Προχωράμε καλά σήμερα και γι' αυτό λοιπόν Νομίζω ότι ενδεχομένω